θέμα. Το επόμενο σημείο μέση διάταξη είναι η σύσταση για δεύτερη ανάγνωση από τον κύριο Κρόιτσμαν, Τελωνιακή Επιβολή των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Κρόιτσμαν, για τέσσερα λεπτά. Έχετε το λόγο, κύριε Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχει κέρια σημασία και για την οικονομία και για τους καταναλωτές. Δυστυχώς το εμπόριο με προϊόντα απομίμησης τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς. Δεν πρόκειται μόνο για προϊόντα πολυτελείας, αλλά και για προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως προϊόντα για τη φροντίδα του σώματος, φάρμακα, παιχνίδια και ηλεκτρικές συσκευές. Όλο και πιο συχνά οι καταναλωτές παραγγέλουν αυτά τα προϊόντα απομίμησης από το διαδίκτυο. Επίσης, τα κυκλώματα των των πειρατικών εμπορευμάτων βρίσκουν συνεχώς νέα μέσα και τρόπους για να μπορούν να ξεφεύγουν από τους ελέγχους των τελωνίων. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί απειλή για τις επιχειρήσεις και για τις θέσεις εργασίας των πολιτών μας. Και πλανούνται οι καταναλωτές και υπάρχουν και κίνδυνοι για την υγεία και για την ασφάλεια των καταναλωτών. Οι εξελίξεις αυτές κατέστησαν απαραίτητη μια επανεξέταση του κανονισμού του 2004 που εξετάζει τη διαδικασία κατάσχεσης και καταστροφής παραποιημένων εμπορευμάτων από τις τελωνιακές αρχές. Οι τελωνιακές αρχές είναι οι ενδεδειγμένες αρχές να αναλάβουν αυτό το έργο γιατί μπορούν να σταματήσουν την αποστολή εμπορευμάτων πριν κυκλοφορήσουν στην εσωτερική αγορά και μοιραστούν σε μικρότερες παρτίδες οπότε θα είναι πιο δύσκολο να, να τα παρακολουθήσουμε. Μετά την πρώτη ανάγνωση πριν από ένα χρόνο περίπου, το Δεκέμβριο του 2012 κάναμε τον τριμερή διάλογο με το, με το Συμβούλιο καταλήξαμε σε ένα κοινό κείμενο. Η Επιτροπή Εσωτερική Αγορά ε, ε, ενέκρινε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ε, με πλειοψηφία 32 υπέρ και 3 ψήφων κατά. Επειδή το Συμβούλιο στι 11 Μαρτίου ήδη ψήφισε τον κανονισμό αυτό, τώρα πρέπει το Κοινοβούλιο αύριο να ψηφίσει επίση τον κανονισμό αυτό για να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία από 1η Πρώτου 2014. Προσπάθησα να επιτύχω δύο στόχου με την έκθεσή μου. Καταρχήν, η προστασία τη πνευματική ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, να απαλλαγούν οι τελωνιακέ αρχέ από τη γραφειοκρατία. Μέσα στον κανονισμό αυτό, οι διατάξει πρέπει να είναι και αποτελεσματικέ και αποδοτικέ και τους δύο στόχους πιστεύω ότι τους έχουμε επιτύχει. Κατορθώσαμε να έχουμε μια πλουστευμένη διαδικασία για την καταστροφή παραποιημένων εμπορευμάτων και αυτό να είναι υποχρεωτικό σε όλα τα κράτη-μέλη και αυτό να επεκτείνεται σε, όλα, σε όλους τους τομείς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να αντιμετωπίσουμε και τις αυξημένες αγορές μέσω διαδικτύου έχουμε και μια ειδική διαδικασία για ε, τις μικρές αποστολές ε, εμπορικού χαρακτήρα. Και εδώ έχει τονίσει τη θέση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα φάρμακα τα οποία βρίσκονται σε διαμετακόμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση φροντίσαμε το τελωνείο να παρεμβαίνει μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένος κίνδυνος να διοχετευθούν στην εσωτερική αγορά. Ε, η ε, τροφοδοσία των ε, αναπτυσσόμενων χωρών με ασφαλή φάρμακα, τα οποία ενδεχομένως παραβιάζουν προστατευόμενα διπλώματα ευρεσιτεχνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται και θα μπορεί μετά την εφαρμογή αυτού του κανονισμού να συνεχίζει να ισχύει. Επίσης, θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με τι ε, τρίτε χώρε για την εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων και αυτό επίση το κατόρθωσε το Κοινοβούλιο με την δουλειά που έχουμε κάνει. Βλέπετε ότι με τα αποτελέσματα λοιπόν ε, τη δουλειά μα είμαστε ικανοποιημένοι. Η έγκριση αυτού του κανονισμού τώρα θα είναι προ όφελο και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και των τελωνιακών αρχών. Ελπίζω ότι αύριο στη ψηφοφορία θα έχουμε την ευρία υποστήριξη του Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και του συναδέλφου και όδη συζητητέ με του οποίου συνεργαστήκαμε θαυμάσια ευχαριστήσω και την Επιτροπή και το Συμβούλιο γιατί πάντοτε ε, είχαμε προτάσεις ε, με τις οποίες μπορούσαμε να δουλέψουμε και πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε όλοι ότι είναι ένας καλός κανονισμός προς όφελος των καταναλωτών και προς όφελος της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κρόιτσμαν και τώρα θα ζητήσω από τον Επίτροπο κύριο Σεμέτα να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΙΜΚΟ και ιδιαίτερα τον εισηγητή, τον κύριο Κρόιτσμαν, για την επικοδομητική προσέγγιση που ακολούθησε κατά τις διαπραγματεύσεις. Η εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τις τελωνιακές αρχές είναι βασική προτεραιότητα της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποτελούν κινητήριο μοχλό της οικονομίας μας και θα πρέπει στους κατόχους των δικαιωμάτων να δίνουμε την βεβαιότητα και ασφάλεια ότι οι καρποί των καινοτομιών τους θα προστατεύονται. Οι τελωνιακές αρχές μπορούν λοιπόν να προστατεύουν αυτό το τομέα και να εμποδίζουν τα προϊόντα πειρατείας να φτάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέληξαν σε συμφωνία για ένα νέο κανονισμό ώστε να επιβάλλονται από τις τελωνιακές αρχές τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Θα σας υπενθυμίσω τα ωφέλη που θα έχουμε από τον κανονισμό αυτό. Καταρχήν, επεκτείνουμε το πεδίο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και μπορούν να επιβάλλουν τα δικαιώματα αυτά στα σύνορα. Τα προϊόντα παραποίηση που στέλνονται σε μικρέ αποστολέ οι ιδιώτε καλύπτονται επίση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν εξετάσουμε ε, τις ταχυδρομικές μεταφορές και τις αποστολές μέσω διαδικτύου τα παραποιημένα προϊόντα και προϊόντα απομίμησης που έχουν ε, ένα παραποιημένο εμπορικό σήμα επίσης καλύπτονται. Αυτό θα κρατήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει το προβάδισμα στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στα σύνορά τη. Δεύτερον υπάρχουν ε, σωστές διαδικασίες ούτε ώστε να έχουμε ένα μόνο αίτημα ε, που θα καλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι απλουστεύεται το έργο των τελωνίων και τηρούνται και τα δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων έχοντας μια διαδικασία χωρίς γραφειοκρατία για όλους τους εμπλεκομένους. Αυτές οι αλλαγές μαζί με τα νέα εργαλεία που δημιουργούνται όπως ε, μια κεντρική βάση, ηλεκτρονική βάση δεδομένων ε, θα, θα κάνει το τελωνίο πιο αποτελεσματικό έναντι των απομιμήσεων και παραποίησεων. Αντιμετωπίζουμε και συγκεκριμένα προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν όσον αφορά την πρόσβαση σε φάρμακα. Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, αλλά έχω την πεποίθηση ότι ε, τώρα το έχουμε ρυθμίσει πλέον οριστικά. Κλείνοντα, ε, η σημερινή συμφωνία θα ενδυναμώσει το νομικό πλαίσιο και θα πλουστεύσει την ε, διοικητική διαδικασία για την κέρια δουλειά που κάνει το Τελωνίο για να προστατεύσει τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. Θα βοηθήσει να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των ε, εμπορευομένων, θα προστατεύσει την ανταγωνιστικότητα τη οικονομία μα που βασίζεται όλο και περισσότερο στην καινοτομία και στην πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό ο νέο κανονισμό είναι καλός όχι μόνο για το τελωνείο, είναι καλό και για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Χάντσλικ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι παραποιήσεις ε, αποτελούν τεράστια απώλεια, τεράστια ζημιά στην εσωτερική αγορά και επηρεάζονται περισσότερο οι κατασκευαστές των οποίων τα προϊόντα παραποιούνται αλλά και οι καταναλωτές οι οποίοι απειλούνται από, λόγω της έλλειψης ασφάλειας αυτών των προϊόντων. Οι παραποιήσεις αφορούν ρούχα αλλά και φάρμακα. Είναι προϊόντα τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό χρειάζεται να παρακολουθούμε στενά τα σύνορα. Μόνο οι τελωνιακοί στα σύνορα μπορούν να είναι αποτελεσματικοί στη δέσμευση και δίμευση αυτών των προϊόντων. Χρειάζεται όμω να έχουν τα κατάλληλα νομικά μέσα στη διάθεσή του. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, ε, τα μέτρα αυτά γίνονται πιο αποτελεσματικά, απλοποιούνται οι δραστηριότητε και ε, τόσο οι δικαιούχοι όσο και οι καταναλωτέ ε, θα είναι περισσότερο προστατευμένοι. Επιπλέον, δεν αλλάζει τίποτα στη διανοητική ιδιοκτησία και δεν επηρεάζονται τα εμπορικά προϊόντα τα οποία φέρνουν οι τουρίστες στις αποσκευές τους ο έλεγχος εκ μέρους των τελωνιακών αρχών ε, θα εφαρμόζει τις ε, διάφορες διατάξεις, νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς αυτές ε, θα είχαμε ένα κενό το οποίο θα οδηγούσε σε τεράστιες ζημίες. Μιλούμε για ζημίες που ανέρχονται περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δεν πρόκειται για μικρό ποσό. Ή τα προσόντα των τελωνιακών υπαλλήλων είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος για δύο λεπτά ε, στην κυρία Χέντ. Ευχαριστώ. Πριν από ένα χρόνο είδαμε με σαφήνεια τα προβλήματα των, ε, της νομοθεσίας μας ε, και το, τώρα όμως ο διάλογος έχει προχωρήσει πολύ, χαίρομαι για το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια νέα νομοθεσία. η οποία θα βοηθούσε πάρα πολύ να μην χάνονται και πολλές θέσεις εργασίας. Ε, δεν είναι μόνο δηλαδή η οικονομική ζημία, αλλά και η ζημία υπό τη μορφή ανεργίας. Ε, πολύ δε περισσότερο που ορισμένα αυτά τα προϊόντα μπορούν να βλάψουν και την υγεία μας. Αυτό που μας ενισχύει είναι να μην διακοπεί η εμπορία και η διακίνηση προϊόντων τα οποία θα θέλαμε να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα φάρμακα. Γνωρίζουμε ότι ορισμένα φάρμακα, γενώσιμα κυρίως, περνούν μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάνε σε άλλες χώρες. Αυτό δεν θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει η Κομισιόν να προστατεύσει αυτές τις, ε, αυτή τη διακίνηση. Και μετά σε μερικά χρόνια θα πρέπει να δούμε μήπως χρειάζεται να προσαρμόσουμε περισσότερο ε, τον κανονισμό αυτό. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ε, μπορούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί περισσότερο και στο μέλλον ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια προθεσμία 10 ημερών για ε, απάντηση και για την ε, προσφυγή στο Δικαστήριο Μικροδιαφορών. Είναι πολύ μικρή αυτή η προθεσμία και λυπάμαι πολύ γιατί καταργείται στην πράξη το δικαίωμα αυτό. Ε, υποστηρίζουμε πάντω τη δεύτερη ανάγνωση, σε δεύτερη ανάγνωση αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπιελάν έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κρόιτσμαν για την έκθεση αυτή που είναι ένα βήμα προς ε, μια πιο αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που θα εξασφαλίσουν ε, τα δικαιώματα των δημιουργών και των καταναλωτών. Τη δημιουργία του νομικού ε, πλαισίου θα εξασφαλίσει ποιοτικά προϊόντα. Υπάρχει ανάγκη αύξηση της προστασίας των ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πράγμα το οποίο υποστηρίζει και αυτή η έκθεση. Ε, όλο και περισσότερες παρτίδες εμπορευμάτων ε, υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα αυτά. Παραποιημένα προϊόντα, προϊόντα απομίμησης που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταφράζονται σε ανεργία. Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι τα παραποιημένα ε, φαρμακευτικά ε, προϊόντα, που είναι το 1 τέταρτο όλων των ε, ε, προϊόντων απομίμησης. Επίσης, μεγάλος κίνδυνος για την υγεία είναι τα παραποιημένα τρόφιμα ή καλλιντικά προϊόντα οι τελωνιακές υπηρεσίες που έχουν περιορισμένους πόρους δεν θα πρέπει να επιφορτιστούν με όλες αυτές τις ε, αρμοδιότητες. Ε, θα πρέπει να αποφασίζεται αν, έχουν ε, καταπατηθεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με βάση την εθνική νομοθεσία. υπάρχουν τεχνολογικές μέθοδοι που μπορούν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο αυτό και χαίρομαι που το δέχεται αυτό το Συμβούλιο. Κυρία Γκάλ Μπέλτς, λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Σιγητά, κύριε Κρόιτσμεν, η διανοητική ιδιοκτησία ε, είναι κέρια σημασία για την ανταγωνιστικότητά μα στην Ευρώπη. Και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία σημαίνει προστασία τη καινοτομία και προστασία των θέσεων εργασία. Η παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα παραποιημένα εμπορεύματα, τα προϊόντα πειρατείας θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να αποτελέσουν πραγματική απειλή για την υγεία των καταναλωτών. Θα πρέπει να προσέξουμε όμως παράλληλα να να, και την δίπτωση που μπορεί να έχουν τα τελωνία. Τέτοιοι κανονισμοί δεν θα πρέπει να επιβάλλουν περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο. Ο κανονισμός αυτός συμφωνεί με άλλους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα ε, πνευματικής ιδιοκτησίας, ε, ενισχύοντας ε, τις τελωνιακές διατάξεις και παράλληλα εμποδίζουμε και τα εμπορεύματα να φτάσουν, τα παραποιημένα εμπορεύματα να φτάσουν στην εσωτερική αγορά. Μπορούν να κρατηθούν στα τελωνία. Οι διαδικασίες αυτές δεν είναι πάντοτε απλές, θα πρέπει να, να τις κρατήσουμε στο δυνατόν απλούστερες. Χαίρομαι γιατί έχει διατυπωθεί αυτός ο κανονισμός με αυτή τη μορφή και υποστηρίζω αυτή την πρόταση κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό, κυρία Κέμπερτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά και τους καταναλωτές και καταναλώτριες, διότι πρόκειται για την ασφάλειά τους και για την υγεία τους. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και θα ήθελα να τονίσω ένα σημείο συγκεκριμένα, τα φαρμακευτικά προϊόντα. Όταν βλέπουμε ότι ένα τέταρτο των κατασχεθέντων παραποιημένων προϊόντων είναι φαρμακευτικά προϊόντα, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι ακριβώς σε αυτό το τομέα να προχωρήσουμε με αυστηρά μέτρα και να μην επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να κυκλοφορήσουν τέτοια προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει ταυτόχρονα να φροντίζουμε μέσω μιας ενδεχομένως κακής διατύπωσης να μην παρεμποδίζεται η διαμετακόμιση γενώσιμων φαρμάκων και να μην προκαλέσουμε, εμείς οι σοσιαλδημοκράτες δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να παρεμποδίσουμε τη διαμετακόμιση τέτοιων φαρμακευτικών προϊόντων από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1,5 λεπτό κύριο Στολογιάννη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους τους αδέλφους που εργάστηκαν για αυτό το κείμενο. Η πρόοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης, η οποία βασίζεται σε μια ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής διανοητικής ιδιοκτησίας. Έχουμε δύο θέματα. Αφενός, έχουμε την νομοθεσία προστασίας τη δυναμική ιδιοκτησία στα κράτη-μέλη, που διαφέρει από χώρα σε χώρα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τις εναρμονίσουμε και από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το γεγονός ότι στις αγορές μας εντοπίζουμε πολλά πειρατικά παραποιημένα προϊόντα, προϊόντα μαϊμού και εκεί θα πρέπει να παρέμβουν οι τελωνιακές αρχές έτσι ώστε να λήξει αυτό το φαινόμενο. Αυτοί που καταδικάζονται για εισαγωγή παραποιημένων προϊόντων πρέπει να υφίστανται τις συνέπειες αυτής της πράξης. Ευχαριστώ. Περνάμε στην διαδικασία Catch the Eye. Καταρχήν ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Ε, ε, Θα ήθελα να συγχαρώ την Κομισιόν και τον εισηγητή για τις ε, τροπολογίες που εισήγαγε. Όλοι οι τύποι παράνομου εμπορίου κοστίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά κατέτος 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι οι προτάσεις αυτές ε, είναι πρακτικές, είναι εφικτό να εφαρμοστούν. Ε, είναι λογικό, δεδομένου τα περισσότερα τέτοιου είδους προϊόντα ε, ότι έρχονται από τρίτες χώρες, είναι λογικό να προσπαθήσουμε να τα σταματήσουμε στα σύνορα. Έχω μία ερώτηση προς τον Επίτροπο πόσα πιστεύετε ότι ε, θα εξοικονομήσουμε από αυτά τα οποία ζημιωνόμαστε αυτή τη στιγμή με τα καινούργια μέτρα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριε Μπέντεργκαστ. Όπως γνωρίζετε η ομάδα μας είχε εκφράσει σημαντικές ανησυχίες στην πρώτη ανάγνωση για αυτό το κείμενο και θέλησαμε πολεμήσαμε για να εξαιρεθούν τα εμπορικά είδη τα οποία φέρουν οι επιβάτες ε, στα ταξίδια τους ε, καθώς επίσης και να εισάγουμε μια απλοποιημένη διαδικασία καταστροφής για μικρές ποσότητες. Ε, χρειάζεται όμως ψηφίσαμε εναντίον της πρότασης διότι θεωρήσαμε στην πρώτη ανάγνωση ότι Επλέτεται η δυνατότητα ε, διαμετακόμισης φαρμάκων μεταξύ τρίτων χωρών. Ε, όμως, στην τροποποίηση που έγινε, ε, βελτιώθηκαν και τα τρία αυτά σημεία ε, έγινε ε, πρόοδος και στο χρονικό διάστημα για την ε, καταστροφή. Αποκλείστηκαν τα προϊόντα που φέρουν οι επιβάτες και διευκολύνθηκε η διαμετακόμιση εμπορευμάτων κυρίως φαρμάκου μεταξύ τρίτων χωρών. Συνεπώς είμαστε ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ. Η κυρία Άντες Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε κύριοι, η κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά αυτή τη στιγμή είναι τέτοια που ε, ένας μικρός αριθμός εμπόρων μπορούν να επιβάλλουν ε, ε προσωρινά μέτρα για ε, στρέβλωση όλης της κατάστασης στην αγορά. Ε, αυτό αφορά ε, όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Αυτό μπορεί να ε, προσπαθήσουμε να το λύσουμε με το σύστημα της, ε, του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Τώρα εφαρμόζουμε νέα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά το θέμα των προσωρινών μέτρων παραμένει ανεπίλητο. Παραδείγματο χάρη ναι, στην αυτοκινητοβιχανία, ξέρουμε ότι οι κατασκευαστέ πολεμάνε με του κατασκευαστές ανταλλακτικών για πολλά χρόνια. Επίσης πρέπει να θεωρήσουμε το παγκόσμιο πρόβλημα. Γιατί ε, ε δεν ε, ε, βλέπουμε το πρόβλημα της Νέας Ιρλανδίας. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι μια αγορά για όλους, ιδιαίτερα για τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εσάια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ ε, τον εισηγητή και τους χιώδης εισηγητές για την πολύ καλή δουλειά τους και την καλή συνεργασία τους με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Χρειαζόμαστε νέους κανόνες στον τομέα αυτό, αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ικανότητα των αρχών μας να κάνουν τη δουλειά τους. η βιομηχανία μας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη απέναντι στην απειλή των παραποιημένων προϊόντων. Είναι προφανές ότι αυτό αποτελεί απειλή και για την υγεία των καταναλωτών μας, ε, ε, δυνάμει τουλάχιστον. Ε, πέραν του οργανωμένου εγκλήματος και του ξεπλήματος ε, ε, χρήματος. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η διαφθορά έχει ένα σημαντικό ρόλο μέσα στο όλο φαινόμενο. Πολλοί από τους καταναλωτές μας όταν αγοράζουν αυτά τα πειρατικά προϊόντα ίσως θα το σκέφτονταν δύο φορές την επόμενη φορά αν ήξεραν τις απειλές για την υγεία τους που σημαίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία η διανοητική ιδιοκτησία αποτελεί παράγοντα ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ε, πνευματική ιδιοκτησία και αυτό στην πηγή. Με την εφαρμογή του άρθρου 50 ε, είμαστε περήφανοι για μια τροπολογία που θεωρούμε σημαντική, που είναι αυτή για την διεθνή συνεργασία όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο, επιχειρησιακό επίπεδο, με την ανταλλαγή πληροφοριών και την υπογραφή συμφωνιών ανάμεσα στις χώρες, το, τους κλάδους και τα τελωνία. Είναι πολύ σημαντική η ε, συνεισφορά της Επιτροπής ίντα μέσω του άρθρου 50. Ωραία. Ο λόγος τώρα στον Επιτρόπο, κ. Σεμέτα. Thank Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ε, απόψεις που εκφράσατε. Αύριο θα ψηφίσετε τον κανονισμό. Με αυτόν τον κανονισμό προσπαθούμε να θέσουμε τις ε, προδιαγραφές παγκοσμίω για αυτό το θέμα. Η ε, αξιοπιστία των θεσμών μας εξαρτάται από αυτό τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις καθορίζονται σαφώς στον κοινωνικό κανονισμό. Νομίζω ότι βρήκαμε και τη σωστή διατύπωση για τα φάρμακα. Είναι πολύ σαφές πια το κείμενο οι κανόνες για το πώς θα χειριζόμαστε τα φάρμακα στα τελωνία. Ο κ. Κέλλη ρώτησε πόσο θα εξοικονομήσουμε με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Λαμβάνοντα υπόψη ότι διευρύναμε το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού, ότι καθορίσαμε σαφεί κανόνε για του τελωνιακού υπαλλήλου και σαφεί διαδικασίε για του δικαιούχου των δικαιωμάτων, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε σημαντικά ποσά. Κάθε χρόνο υποβάλλουμε έκθεση με συγκεκριμένα νούμερα για τα ε, ε, παραπημένα προϊόντα τα οποία ε, δημεύουμε στα σύνορα, θα είναι πολύ εύκολο να ε, παρακολουθήσουμε το πόσο θα ακριβώς εξοικονομούμε. Τα κράτη-μέλη από την άλλη μεριά θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτόν τον κανονισμό. Η Κομισιόν θα υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία συμπεριλαμβανομένου και μέσω της ε, κατάλληλη υποδομή ανταλλαγή πληροφοριών. Περιμένω μια θετική ψήφο από εσά. Ευχαριστώ. And the last is Ευχαριστώ και πάλι ο λόγος στον κύριο Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να τονίσω ότι ποτέ δεν συμπεριλάβαμε τον τουρισμό στον κανονισμό αυτό και η μεταφορά γενώσιμων φαρμάκων επίσης ε, έχει εξαιρεθεί και δεν ε, υπάρχει πρόβλημα με φάρμακα για τον τρίτο κόσμο. Και χαιρόμαστε για τον κανονισμό αυτό που έχει φτάσει στο Κοινοβούλιο. Είναι τεράστια σημασία ε, η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό σημαίνει θέσει εργασία. Είναι σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για του καταναλωτέ, όχι μόνο για τι επιχειρήσει, αλλά και για του καταναλωτέ. Ε, ε, έχω δει τρομακτικέ εικόνε, ε, γιατί άνθρωποι έχασαν τα δόντια τους γιατί πήραν κάποια φάρμακα τα οποία ήταν απομιμήσεις φαρμάκων. Καταρθώσαμε να συμπεριλάβουμε τρία στοιχεία σε αυτόν τον κανονισμό. Να μειώσουμε τη γραφειοκρατία στα τελωνία για να δουλεύουν πιο αποτελεσματικά τα τελωνία και αυτό το επιτύχαμε μέσω τη απλουστευμένη διαδικασία, γιατί μπορεί και πάλι το τελωνίο να μην χρειάζεται δικαστική διαδικασία μετά από την αίτηση του ε, ε, δικαιούχου των δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα, τα δικαιώματα των ε, ε, δικαιούχων τα έχουμε ενισχύσει και αυτό το έχουμε επιτύχει με αυτόν τον κανονισμό και στο μέλλον θα μπορεί ε, ο δικαιούχος να αποζημιωθεί για την καταστροφή από τον, αυτόν που έκανε την παραποίηση. Και το τρίτο είναι επίσης προστασία των δεδομένων και αυτό θέλω να το τονίσω γιατί η προστασία των δεδομένων επίση είναι πολύ σημαντική όταν χειριζόμαστε τέτοια θέματα και την έχουμε ενισχύσει την ε, προστασία των δεδομένων. Πιστεύω ότι ε, με την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο βελτιώσαμε ακόμη περισσότερο την καλή πρόταση τη επιτροπή και ελπίζω αύριο θα έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία. Είναι μια συμβασική λύση που ελπίζουμε ότι θα

ψηφιστεί ούτως ώστε από 1η Πρώτου 2014 να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμό. Και είναι και σημαντικό επίση οι εθνικέ τελωνιακέ αρχέ να έχουν αρκετό προσωπικό στη διάθεσή του στην χώρα μου, στη Γερμανία. Λείπουν 8.000 ε, τελωνιακοί. Η Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει ε, να φροντίσει, να, να πιέσει και σε εθνικό επίπεδο να δοθούν οι κατάλληλοι πόροι στις υπηρεσίες αυτές Πιστεύω ότι θα αποτελέσει πρόοδο για τους καταναλωτές, για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και για την ενδυνάμωση των προτύπων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Κρόιτσμαν. Πέρα τη συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30. Κυρίε και κύριοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η